ότι εξ ονόματος ε, Πολωνού ε, δικηγόρου θέλουμε να ζητήθηκε να αρθεί η ασυλία ενός συναδέλφου του Κοινοβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 3 της, ε, του κανονισμού οι εντολές του κυρίου Αγκουράκη, Στανέλης και Σαραβράκος ελέγχθησαν